στις 8 ε, ε, Φεβρουαρίου. Θα ήθελα καταρχήν ε, να καλωσορίσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Χέρμαν Βαρόπο, για πρώτη φορά στην παρθενική του εμφάνιση στην Ολομέλεια. Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να προθερμαθούμε και να ξεκινήσουμε στη συζήτηση. Κανένα 15 λεπτό για τα δικαστικά. Θα ήθελα επίση να καλωσορίσω θερμά και τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Μπαρόζο, που είναι συνήθι γνώριμο στι τελευταίε πενταετίε. Δεν είναι καινούρια λοιπόν η παρουσία του κύριου Μπαρόζο στην ολομέλειά μα. Και θα ήθελα στην αρχή να κάνω ορισμένε παρατηρήσει, αγαπητοί συνάδελφοι. Με θλίψη καταρχήν θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρα κοντά στις Βρυξέλλες έχασε τη ζωή της και η κυρία Κλάουδια Καντεάγκο